Dear colleagues, welcome to IMCO. Συνάδελφοι, καλώ ήρθατε. ξεκινήσουμε αρχικά με την εξέτηση τη μέσα διάταξη Να σα πω ότι η ψηφοφορία για τι ε, εταιρείε περιορισμένη ευθύνη έχει αναβληθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια για τη μέσα διάταξη, αλλιώ θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί και προχωρούμε. Ανακοινώσει ε, του Προέδρου. Δεν έχουμε τελική απόφαση για την DSM, την έκθεση που έχει ζητήσει η ΊΝΚΟ. Υπάρχουν ζητήματα για την προστασία καταναλωτών και πραγματικά πρέπει και η Επιτροπή μας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην DSM, σε συνεργασία και μάλιστα επιτροπές που τον κανόνα 55, 54 μάλλον, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε. Ενθυμίζω ότι μεταδίδεται μέσω διαδικτύου η συνεδρίαση αυτή. Καλώ ορίζουμε όσοι την παρακολουθούν. Εφαρμογή e-meeting. Το e-meeting και τα... μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί προ πολιτικέ ομάδε, βοηθή. Α γεννήσουμε λοιπόν εμεί την ψηφιακή Ευρώπη. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το πολύ καλό μας ενημερωτικό δελτίο, το newsletter, υπάρχουν 60 είναι το τεύχος αυτό, είναι στη διάθεσή σας. Και όσοι θέλετε μπορείτε να το λαμβάνετε και συστηματικά, αν θέλετε να παρακολουθείτε τις εργασίες μας. Τώρα περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 22ης Ιουνίου. Θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί λοιπόν. Και τώρα ας περάσουμε στην ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο. Έχουμε την έκθεση ε, για τις εγκαταστάσεις ε, καλωδίων, ψηφιστικές ε, εγκαταστάσεις και εφαρμογές. Ο κύριος Λόπες είναι εδώ μαζί μας. Θέλει να μας πει δύο λόγια. Thank you, President. Um, I will turn to Spanish. Συνάλφη, στις 11 Ιουνίου έλαβε χώρα η, η, η τελευταία συνάντηση του τριμερούς ε, διαλόγου μετά από δύο-τρεις πρώτες τεχνικές συναντήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ε, εργαστήκαμε από κοινού όλες οι ομάδες, κάτι που έδειξε ότι η Επιτροπή μας ενωμένη, είναι ενωμένη και παρούσα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την πρόεδρο της Επιτροπής μας για τον ρόλο που έπαιξε κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων. Τέσσερα σημεία θέλω να υπογραμμίσω. Τέσσερις επιτυχίες θα έλεγα αυτών των διαπραγματεύσεων. Πρώτον, ε, περισσότερη πληροφορία για τους καταναλωτές, ε, με μεγαλύτερη αναφορά των παραγωγών ε, στα site, άρθρο για το θέμα του της ε, του, της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας. Τρίτον, ε, ένα άρθρο πιο πλήρες για τις κυρώσεις και μια καινούργια παράγραφο της εταιρολικής έκθεσης. ενισχύσαμε το σύστημα κυρώσεων του κανονισμού με τους πιο εισηγητές. Τέταρτον, διορθώσαμε το, τα όσα αναφέρονταν σε ό,τι αφορά τις ε, παλαιότερες εγκαταστάσεις, ιστορικές εγκαταστάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Εκεί θα έχουμε μια ξεχωριστή κατηγορία ε, ε, εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986, δηλαδή έχουν ηλικία πάνω από 30 έτη. Τα, οι υπόλοιπε εγκατα... ιστορικέ εγκαταστάσει μπορούν να θεωρηθούν ε, ω ε, εγκαταστάσει ενδιαφέροντο, αλλά θα πρέπει να λάβουν τι κατάλληλε ε, τεχνικέ εγκρίσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Λούση Άντερσον και του υπόλοιπου σκιώδει ηγητέ και όλου όσου εργάστηκαν, συνεργάστηκαν, του συμβούλου μα, ε, την Άστριτ και τον Σεβαστιάν. Νομίζω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ. αυτό το θέμα ήταν τεχνικά και τεχνολογικά πολύ περίπλοκο εξ αρχής, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε και με επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τον κύριο Αντώνιο Λόπες. Τώρα, συνάδελφε, είσαι εισηγητής ε, για τις ε, συσκευέ του Σκοερίου. Δεν ξέρω αν θέλετε να επέμβετε. Ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κοινή συνεδρίαση για τον προσταστικό εξοπλισμό και τις ε, καταστάσεις του Σικοαρίου. Είχαμε εκτενείς ε, συζητήσεις για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι σημειώνεται πρόοδος στο πρώτο ζήτημα του προσταστικού εξοπλισμού. Ακόμα εκρεμούν κάποια ζητήματα. Δεν είμαι εισηγήτρια βεβαίω, απλώ είμαι επικεφαλή του διαλόγου και ελπίζουμε ότι θα ε, βρεθούν λύσεις για τον εξοπλισμό φυσικού αερίου που είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο ζήτημα αλλά ακόμα κάποια συστήματα πρέπει να βελτιωθούν. Έχει σημειωθεί ο πρώτος και αν δεν κάνω λάθος νομίζω θα περάσει στην Προεδρία του Λουξεμβούργου και νομίζω θα, το εξετάσουμε και την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος κύριε Πρόεδρε, αλλά ελπίζουμε να το λύσουμε ζήτημα, να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα και στους δύο αυτούς τομεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, άλλα σχόλια για τον τριμερή διάλογο. Όχι. Εισηγητή για το επόμενο θέμα για την γνωμοδότηση για, τις, ε, για του κινητήρε εσωτερικής καύση που προορίζονται για μειωδικά κινητά μηχανήματα δεν είναι εδώ η εισηγήτρια, επομένω να την περιμένουμε. Α ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο. Α, και στο επόμενο είναι η εισηγήτρια όμω. Okay. Ας περάσουμε λοιπόν στην πρώτη γνωμοδότηση. Ανδρέας, δεν ξέρω, θες να πεις δύο λόγια εξ ονόματος της συζητήτρες ε, του ΕΠΠ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω δύο λόγια ως ε, ε δεδομένου του εισηγητής του επόμενου θέματος δεν είναι παρόν να πω δύο λόγια για τον τριμερή διάλογο για την ασφάλεια των ε, δικτύων. Ε, αν μιλήσω υπερβολικά πολύ και μακρηγορήσω και φτάσει η πέστε μου κύριε Πρόεδρε. Να ενημερώσω αγαπητή κυρία Πρόεδρε τους ε, συναδέλφους ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε εκ νέου με τους κοιόδες ε, εισηγητές και συμφωνήσαμε ότι δεδομένου των πολλαπλών κινδύνων και των πολλαπλών κυβερνεπιθέσεων ε, εις βάρος των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όπως η πολωνική ΛΟΤ σήμερα εκ νέου, δεν θα πρέπει να επαναχωρήσουμε σε σχέση με αυτά που ψηφίστηκαν στο, στην προηγούμενη θητεία στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξοπλιστούμε με την απαραίτητη υπομονή. Να ευχαριστήσω και τους κοιόδης ε, γιατί θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με τον σωστό τρόπο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Με ενιαίο νομικό πλαίσιο. Για να διασφαλίσουμε ότι σε λίγους μήνες σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει μία άμυνα, σε ό,τι αφορά τις κριτικές υποδομές, παρούμια, ίσου επίπεδου. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Και το θέμα της αλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, το ερώτημα του πώς ε, θα συμπεριληφθούν και πώς θα οριστεί το πεδίο εφαρμογή ε, της νομοθεσίας, αλλά το βασικό είναι να προστατευτεί οι κρίσιμες υποδομές σε ό,τι αφορά και την οδηγία και τι προβλέπεται. Η ηλεκτρονική προεδρία ε, είναι πολύ υποκατομητική στις διαπραγματεύσεις της, γι' αυτό ελπίζουμε να πετύχουμε τουλάχιστον μια πρώτη πολιτική νίκη, ακόμα και αν δεν καταλήξουμε σε κάποιο οριστικό και ολοκληρωτικό αποτέλεσμα στον τριμερή διάλογο της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ για την κυβερνοασφάλεια, για την ενημέρωση αυτή, για την ασφάλεια, για τα όρια ρήπων για τα οδικά οχήματα θα θέλετε. Μήπως να μιλήσετε εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ο κ. Φανίστηλ θα να μιλήσει και δεν τον βλέπω. Αλλά μπορώ γρήγορα γρήγορα να ελέγξω και να ψάξω να δω που είναι. Η πρόεδρος. Ας δώσουμε λοιπόν τότε το λόγο κατευθείαν στην σκιώδη εισηγήτρια την κυρία Γκραπίνη. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι εξετάζουμε τις 35 τροπολογίε που έχουν κατατεθεί για το σχέδιο γραμματότητα. Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής δεν είναι εδώ, αλλά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον εισηγητή και με τους κοιόδης εισηγητές. Έγιναν πολλές συναντήσεις και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες με τι ε, συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες πετύχαμε, νομίζω καταλήγουμε σε μια συνέντευξη και νομίζω ότι πλέον είναι πολύ στεναρή η γνωματοδότηση, η οποία είναι πάρα πολύ τεχνική φύσεως, αλλά πάρα πολύ σημαντική κιόλα. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί καταρχά αφορά θέμα ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά, αλλά πέραν αυτού άπτεται και θέματα προστασία του καταναλωτή. Πιστεύω λοιπόν ότι με τις τροπολογίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και για τον εξοπλισμό και για τα μηχανήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια παρόμοια ποιότητα και ίσης, ίσα πρότυπα προστασίας να υπάρχει και η σωστή τεκμηρίωση, αλλά εκ παραλλήλου να φροντίσουμε μέσω το, της μη ελεγχόμενης εισαγωγής να μην καταλήξουμε σε εισαγωγή προϊόντων που θα υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ένα σωστό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές για να προστατεύσουμε το καταναλωτή από ατυχήματα αλλά και το περιβάλλον από μόλυνση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εκ νέου τον εισηγητή και τους κοιόδης για την πολύ ευχάριστη συνεργασία και ελπίζουμε με τον τρόπο έτσι να συμβάλλουμε στην ε, έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και επίσης να είναι μια έκθεση αυτή με πρακτική συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ Μαρία από το ECR. Ε, Θα επαναλάβω και εγώ αυτά που είπε η κυρία Γκραπίνη. Δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ε, ο συμβασμό είναι πολύ θετικός. Από τη δική μας πλευρά χαίρομαι που η τροπολογία μου υπαριθμών 48 που επέτρεπε τους κινητές αντικατάστασης ε, που έχουν παραχθεί πριν από τον Ιανουάριο 2011 να μπορούν να τύχουν εμπορίας, να τεθούν σε εμπορία. Ε, χαίρομαι που πέρασε. και θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή και τους άλλους και εισηγητές σε ό,τι αφορά και την μεταβατική περίοδο για την αντικατάσταση των κινητήρων. Νομίζω ότι ο συμβασμός είναι πολύ καλός. 18 μήνες πλέον η μεταβατική περίοδος. αλλά λαμβάνονται υπόψη και ισχύοντες ε, κανόνες ε, ε, κρατικών προμηθειών και ισχύοντες κανονισμοί και προκειμένου να λειτουργήσει αυτό ο συνδυασμός θέλω στην παριθμό 19 τροπολογία να πούμε με ε, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2008-57 και του κανονισμού 1302 του 2014 προκειμένου ε, αυτό προτείνω να προσθεθεί στην τροπολογία παριθμών 19 για να λειτουργήσει ο συμβασμός. Όμως ο, η συμφωνία έχει επιτευχθεί, η ομάδα μου είναι ικανοποιημένη και μπορώ να την υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων τώρα. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to apologize, η κυρία Τσαρντζόβα. Θα ε, σας παρουσιάσω εγώ μια σύνοψη της άποψής μας. Οι συζητήσεις ήταν πολύ καλές. Ο εισηγητής ε, ε, βοήθησε πολύ στο να ανεβρεθεί μια ισορροπία. Κανοποίηθηκαμε σε ό,τι αφορά και τη μεταβατική περίοδο και σε ό,τι αφορά τους ε, κινητές αντικατάστασης. Ε, γιατί αυτές ήταν οι ανησυχίες μας αρχικά. Τώρα μπορούμε να υποστηρίξουμε το συμβασμό εκ λοιπόν των φιλελευθέρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους άλλους πιο εισηγητές για την καλή συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος, άλλα σχόλια από άλλους συναδέλφους, άλλες πολιτικές ομάδες. Ωραία. Δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχη αυτή η γνωμοδότηση λοιπόν. Θα ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα στις 23 Ιουνίου στην Επιτροπή μας η Επιτροπή ΕΜΒΗ θα ψηφίσει στις 15 και 16 Ιουλίου και στην Ολομέλεια, δεν ξέρουμε σε ποια Ολομέλεια, πότε θα ψηφιστεί, εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην έκθεση πρωτοβουλία. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μιλήσουν τώρα. Ε, έκθεση πρωτοβουλία. Ε, ο εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς εισηγητή ο κ. Σουβάμπ. Ε, βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασία των τροπολογιών. 67 συγκεκριμένε τροπολογίε έχουν υποβληθεί. Μαρία, θες να πάει στο λόγο, να ξεκινήσεις εσύ, εκ μέρου των σοσιαλιστών. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντω. Νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί ήταν εξαιρετική η συνεργασία με τον Ανδρέα Σβάμπ και πρόκειται για μία έκθεση με καλή δομή, ισόρροπη δομή. Ευχαριστώ λοιπόν τον Ανδρέα και για την ε, πληρότητα του κειμένου. Είναι τόσο πλήρη μάλιστα η έκθεση που δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλέ προσθήκε. Η κοινωνική ωστόσο διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα μου και κυρίως σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε τις σχετικές συμφωνίες με την Ελβετία. Και για το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι σε ό,τι αφορά θέματα αμοιβαιότητα ε, μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΕΟΧ. Ως κοιόδης λοιπόν ε, εισηγητρία πρέπει να σα πω ότι δεν αντιμετώπισα προβλήματα με την έκθεση ούτε με τον εισηγητή. Αλλά η τροπολογία υπαριθμού 4 ότι η Ελβετία θα πρέπει να πληρεί τι ε, απαιτήσει που πηγάζουν από την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι η δράση αυτή και μάλιστα αν δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η Ελβετία, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό υποδεικνύουμε ακριβώς αυτή την ε, τροπολογία. Θα ήθελα επίση τροπολογία 6. Να υπογραμμίσω το εξή. Ο τα μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Εξωτερικής Πολιτικής συνεργάστηκαν ιδιαίτερα στον τομέα αυτό για να υπάρξει σωστή ενιαία αγορά. Και είναι λοιπόν καλή συνεργασία πλέον μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά και τις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ. Επίσης, είναι σημαντικό ότι η... είναι σωστή διάσταση στην, ε, στο δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και προστασία των θέσεων εργασία. Και αυτό αποτυπώνεται στην τροπολογία μου υπαριθμό 1. Συνοψίζοντα, θεωρώ ότι η δουλειά του Ανδρέα σε συνδυασμό με τη δουλειά των σκηνοδών θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα καλό προκειμένου και η Ελβετία και ο ΕΟΧ να βελτιωθούν σε ό,τι αφορά τη εργασία μα μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο. Ποιο θα μιλήσει τώρα από το ACR, Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Ντάλτον. Ο κύριο Ντάλτον, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι και ο συνάδελφο ήθελε να πάρει το λόγο αυτό το ζήτημα και λυπούμε που δεν είναι εδώ. Δεν έχω ακριβώ τι σημειώσει του, επομένω δεν μπορώ να πω ποιε είναι ακριβώ οι θέσει του. Να σα πω τη δική, μας, ε, δική μου γνώμη, μάλλον προσωπική. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε και να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο στην Ελβετία, γιατί πήραν την απόφασή του και την, και την εξέφρασαν και ξεκάθαρα. Πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν καταλήξει σε μια ικανοποιητική λύση η Ελβετία ποτέ δεν ήταν πλήρες μέλος ε, της ε, ενία αγοράς και η διμερή συμφωνία μέχρι τώρα είχε συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Ενώ η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερία και πυλώνες της ενίας αγοράς, και τα άτομα αυτά που κινούνται θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, να ζήσουν, να έχουν δηλαδή τα απαραίτητα προ το ζήν. Αυτό είναι και μια απαραίτητη υποχρέωση για την ελεύθερη ε, κίνηση και κυκλοφορία προσώπων. Επίση, θεωρώ θεμελιώδε ζήτημα το ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων θα πρέπει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και στην προσφορά και ζήτηση τη αγορά και στι δεξιότητε που προσφέρονται και στι ευκαιρίε που υπάρχουν στις χώρες υποδοχή. Ιδάλω θα δούμε ένταση των προβλημάτων που βλέπουμε και στην Ελβετία και μα απασχολούν αυτά τα ζητήματα και στον Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μεγάλοι αριθμοί προσώπων έρχονται σε ορισμένε χώρε και ορισμένε φορέ ε, διαταράσσεται η ισορροπία που έχουμε μεταξύ προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασία. λοιπόν να εξετάσουμε με συμπάθεια αν θέλετε και συμπόνια την Ελβετία και όχι να τους αποκλείσουμε επειδή ο ελβετικός λαός πήρε μια απόφαση για το ποιος θα έρχεται στη χώρα τους ε, και ποιος όχι. Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων λοιπόν είναι απαραίτητη ελευθερία, αλλά δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που διέπει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Ευχαριστώ και εξ ονόματος της Άλντε, κυρία Σανάτσοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματο του κυρίου Σατουρνά, θα μιλήσω, της κυρίας Τουρνά, αλλά έχω και κάποιες σημειώσεις από πλευρά τη. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότηση, πολύ καλή βάση περαιτέρω συζητήσεων. Ορισμένε παρατηρήσει για τι τροπολογίε. Συμφωνούμε με τροπολογία 5 απογραμμίζεται η σχέση μεταξύ των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων TTIP στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανών επιπλοκών για τα κράτη-μέλη ε, του ΕΟΧ. Είναι ένα θετικό στοιχείο πρέπει να προσθεθεί. Για την παράγραφο 6 και 7 τα θέματα μεταξύ ε, χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ, ΕΦΤΑ πρέπει να επιληθούν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε και ελπίζει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία εδώ. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες που αλλάζουν το ποσοστό σε ό,τι αφορά το έλλειμμα μετάβασης και ο συγκεκριτής δεν έχει αντίρρηση. Πρέπει μόνο να διορθωθεί. Για τροπολογία 40, επιμέρους προϊόντα, ιδίως στο γεωργικό τομέα, έχει προσέξει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες ε, δυσκολίες με την αύξηση εισαγωγικών δασμών. Κάποια ζητήματα έχουν επιληθεί, αλλά όχι όλα. Γι' αυτό θέλει να παραμείνει η παραπομπή αυτή, όμω αν υπάρχουν ε, ερωτήματα είναι διατεθειμένη να τα εξηγήσει περαιτέρω. Επομένω, να σα μεταφέρω ότι προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και του Σκιώδη. Ευχαριστούμε, Ντίτα. Από τι άλλε πολιτικέ ομάδε υπάρχουν σχόλια. Ο κύριος Διουρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνει το λόγο. Δύο λόγια μόνο. Εμεί δεν καταθέσαμε τροπολογίε, όμω ήθελα αρχικά να υπογραμμίσω ότι το εξαιρετικό έργο του κυρίου Σουάμπ για αυτό το ζήτημα. Και. Εντάξει, δεν θέλω να απαντήσω, απλώ να παρατηρήσω ότι η βούληση για την εξέβρεση ισορροπίας είναι απαραίτητο στοιχείο μεταξύ υποχρεώσεων και καθηκόντων. Ξέρω λοιπόν ότι κάποιοι θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμπνευση, σε ό,τι αφορά, μεγαλύτερο βάρος δηλαδή σε ό,τι αφορά την προτίμηση ε, ενός λαού, αλλά από την άλλη πρέπει να εξετάσουμε και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ε, που προκύπτουν ε, από μια τέτοια συμφωνία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βρούμε και να αναζητήσουμε αυτή την ισορροπία. Ακριβώς αυτό επεδίωξε ο κύριος Σουάμπ και τον ευχαριστώ παρότι δεν ε, βρίσκεται εδώ και τον συγχαίρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι προτρέχουμε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Επομένω, κάποιοι συνάδελφοι που είχαν ε, προγραμματίσει την παρουσία τους. Δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε που δεν βρίσκονται εδώ. Το ίδιο ισχύει και για εσά. Σίγουρα δεν θα τους κατηγορήσει κανείς και θα τους ενημερώσουμε πλήρως για τα όσα συμβαίνουν στην συνάντησή μας. Γιατί να έχετε κι εσείς κατά νου ότι δεν μπορούμε πάντα να τηρούμε κατά γράμμα το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, θα ανοίξει ο κατάλογος ομιλητών. Κύριε Κέπαρτ, παρακαλώ σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πολύ καλή το πολύ καλό σχέδιο, το οποίο δίνει και μια πολύ καλή γραμμή. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα σημείο και να το υπογραμμίσω από πλευρά από τη ομάδα μα, όπω είπε και η Μαρία, αλλά και ο Πασκάλ το έθεσε. Και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Τάλτον στέκει αυτό που είπατε κύριε Ντάλτον, ότι θα πρέπει να σεβόμαστε αυτά που αποφάσισε ο λαός της Ελβετίας. Δεν μπορούμε απλά να τα γνωρίσουμε. Είναι σημαντικά. Ωστόσο, η Ελβετία έχει προσυπογράψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να σεβαστούμε και τις συμφωνίες αυτές και να φροντίσουμε ότι θα γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες σε ό,τι αφορά τα βασικά, τις βασικές θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών λοιπόν συγκαταλέγεται και η ελευθερία κίνησης. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρεις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μερικοί εξ αυτών να μην έχουν ίδια δικαιώματα με κάποιους άλλους. Αυτό δεν σηκώνει ούτε αλλά ούτε όμως ούτε τίποτε άλλο. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε μέσω συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω συμφωνιών με άλλες χώρες, ισχύει για όλους. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα συμβιβασμό που να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ όλα η πρόεδρος, ευχαριστούμε την κυρία Κέφχαρτ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Στάλερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε να ευχαριστήσω και όσου ε, πριν το λόγο. Καταρχά να διευκρινίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η έκθεση μιλάει για τα ε, λύματα ε, μεταφορά σε ό,τι αφορά το scoreboard. Είναι κάτι το οποίο υπογραμμίσαμε και στις συναντήσεις γιατί παρευρέθηκα στις συναντήσεις με τον ΕΟΧ και την ΕΖΕΣ και στην συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω κάποια ζητήματα. Οι Ελβετοί ψήφισαν όντω πριν το προηγούμενο δημοψήφισμα για να υποστηρίξουν τους κανόνες της ιστορικής αγοράς και στη συνέχεια το δημοψήφισμα το Φεβρουαρίο του 2014 ανέτρεψε την ε, απόφαση αυτή. 50,3% είναι το αποτέλεσμα στο στη δημοσκόπηση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό στο δημοψήφισμα, συγγνώμη. Αυτό τι σημαίνει ότι μέχρι το 2017 θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών. 300.000 άτομα ε, καθημερινά ε, μετακινούνται προς την Ελβετία για να δουλέψουν. Τι θα γίνει με τους πολίτες αυτές. 1,3 ε, εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης ζουν στην Ελβετία. Τι θα γίνει λοιπόν όταν περάσει η νομοθεσία αυτή δεν ε, πρόκειται για κάτι αμαλυτέο. Πρόκειται για μια νομοθεσία που θα επηρεάσει πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες που αμα, δούλευαν, πήγαν φόρους στην Ελβετία. Και αυτό λοιπόν εγκρίθηκε από ένα δημοψήφισμα. Εγκρίνεται η νομοθεσία, η νομοθεσία αυτή και μετά γίνεται άλλο ένα άλλο δημοψήφισμα που απορρίπτει το πρώτο δημοψήφισμα. Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε λοιπόν. Ποια θα είναι η μεταχείριση των ατόμων αυτών. Όπως είπαν και άλλοι, αυτό το δημοψήφισμα θα έχει συνέπειε. Και στη συνάντηση που έγινε στη Ζηρική πριν από κάποιες εβδομάδες, σίγουρα λαμβάνεται και λήφθη σοβαρά υπόψη. Είναι σημαντικό όμως να αναφερθούμε όχι μόνο στην Ελβετία, αλλά και στη σκόρμπο της ιστορική αγοράς και το πώ διασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και πιο γρήγορη και πιο σωστή εφαρμογή των οντών για την εσωτερική αγορά. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να θέσω μερικά σημεία, αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Στάιλερ. Κανένα άλλο συνάδελφο θα θέλει να πάρει το λόγο να σχολιάσει. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πάρω εγώ το λόγο λοιπόν τώρα. Ως ε, μέλος της ομάδας του ΕΛΚ θα ήθελα να συμφωνήσω ότι με πολλά από αυτά που υπόθηκαν σίγουρα θα πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προφανώς αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να κάνουμε διακρίσεις βάρος και να γίνονται διακρίσεις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την ελευθερία ε, διακίνησης. Ε, ε, και όπως δεν το δεχόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιου είδου διακρίσεις ε, και σε χώρες ε, εταίρων ή φίλων μας. Ε, ο Ελβετός Πρέσβης ήρθε εδώ συζητήσαμε τις ελβετικέ αρχές, το καταστήσαμε σαφές. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι à la carte, όπου κάποια χώρα να υποφελείται από τα θετικά, όπως ε, την εναρμόνιση εσωτερικής αγορά, ε, την ε, ασφάλεια και τη σταθερότητα κλπ. Και ταυτόχρονα να μην σεβόμαστε όλους τους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν σεβόμενοι τις αποφάσεις του ελβετικού λαού να υποσκάψουμε τη δική μας εσωτερική αγορά. Είναι κοινή μας ευθύνη να να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό και όλες αυτές τις ε, πολιτικές ε, δυνάμεις, τις οποίες δυστυχώς έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι παρούσες μόνο στην Ελβετία. Οπότε θα πρέπει όλοι μαζί από κοινού να εξηγήσουμε, να διευκρινίσουμε και να υποστηρίξουμε ε, την διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Και ελπίζω ότι οι ελβετικές αρχές θα το καταλάβουν. Θέλω να συγχαρώ τον Ανδρέα Σφάπ για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει μια ισορροπία. Το θέμα είναι ιδιαίτερα κανθόδες. Αυτά. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στις 15 Ιουλίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 16 Ιουλίου. Περνάμε στην ε, γνωμοδότηση για τη μείωση των εκπομπών ρήπων από οδικά οχήματα. η συγγήτρια Ρώσα Φοντούν und Χόλενστάιν συζητούμε τις, τις, ε, γνωμοδο, τις ε, τροπολογίες ε, ε, της υπεύθυνη έμβη 75 ε, τροπολογίες έχουν κατατεθεί συμπεριλαμβανομένων 13 στο σχέδιο ε, ε και μία συμβιβαστική τροπολογία έχει συζητηθεί. Ο ο σκιός ηγητής των σοσιαλιστών, η Λένα Άντρουσον, ε, δεν ξέρω αν θέλει κανείς να μιλήσει εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Εύελιν, εκ μέρους των σοσιαλιστών, ωραία. Δεν προβλεπότανε, αλλά... Η κυρία Τούν ε, Χονστάιν ε, και οι συγκεκριμένοι νομίζω έκαναν καλή δουλειά και νομίζω ότι όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για να φροντίσουμε ότι θα βελτιωθεί η οικολογική προστασία. Το πλαίσιο στο οποίο ζει ο άνθρωπος για τη μείωση των εκπομπών, όλα αυτά μόνο θετικά λοιπόν μπορούν να είναι. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και νομίζω ότι οι συμβαστικές προτάσεις που έχουμε πλέον ε, κοιτάπητο αποτελούν καλές προτάσεις με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν θα μπορούσα να πω τίποτα παραπάνω στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Εύελιν. Και τώρα, εξ ονόματος του ECR, θα δώσουμε το λόγο στην Κρεντάλτο να κάνουμε πρώτα τον γύρο των πολιτικών ομάδων και μετά θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Πρώτα πολιτικές ομάδες, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε μου για πίεση. Θα κάνω γρήγορα. Από δική μα πλευρά, ε, Καλωσορίζουμε μια σειρά στοιχείων στον αναφερειμένο κανονισμό σε ό,τι αφορά τη μείωση των επιβαρύνσεων στου παραγωγούς και σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις τη Ευρωπαϊκή. Επιτροπή. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ε, ε, βελτίωση για τους παραγωγού. ιδιαίτερα τι προτάσει για τη μείωση της αμμονίας για την, ε, το μεθάνιο επίση και για ε, ε, την ταξινόμησή του και την χαρακτηρισμό του ως αέριο του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με όλα αυτά. Τώρα, να περάσω στα προβλήματα που είχαμε μεταξύ των σκιωδών. Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσω πράξεων κατά ταξιοδότηση ή μέσω τροποποίηση της βασικής νομοθετικής πράξης και πώς. Από δική μας πλευράς, και εδώ είναι αρκετά στεναρή άποψη της ομάδας μου. Θα θέλαμε. Τα τμήματα του κανονισμού που ορίζουν οριακές τιμές να μεταβάλλονται μέσω συναπόφαση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να το αποφασίζει μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελούν κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα και θα πρέπει να τα αποφασίζουν οι συνομοθέτε. Αυτή είναι η θέση μα. Ωστόσο, για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπω για παράδειγμα τη ελέγχων, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τι ωριακέ τιμέ όμω, τι τιμέ ορίων, αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται μέσω στην απόφαση. Ένα άλλο βασικό θέμα από πλευρά μα είναι οι μετρητέ, ε, οι υποχρεωτικοί μετρητέ κατανάλωση ε, καυσίμων. Δεν υποστηρίζουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα για μια σειρά λόγων. Καταρχάς το κόστος. Πολλοί μου λένε ότι δεν χρειάζεται να κοστίσει αυτό τίποτα, γιατί υπάρχουν ήδη τέτοιοι μετρητέ. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί αν υπάρξει υποχρεωτικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρξουν και τα του προδιαφέ. Που να πληρούνται από όλου του μετρητέ. Άρα θα πρέπει να αλλάξουν τα συστήματα ενδεχομένω για να προσαρμοστούν στι τεχνικέ προδιαγραφέ που θα ορίσουμε. Άρα θα υπάρξει κόστο. Κατά δεύτερον, υπάρχει και ένα πραγματικό θέμα για τους μικρούς παραγωγούς και έχουμε πολλούς στην περιφερειά μου, γιατί δεν βάζουν υπολογιστές ε, στα αυτοκίνητα αυτή η μικρή παραγωγή. Πολύ ανησυχώ λοιπόν για τον αντικτύπο της υποχρεωτικής αυτής της περίληψης μετρητών. Δεν είμαι κατά των μετρητών εν γέννη. Είναι καλή ιδέα πιστεύω για την ε, μέτρηση της καταναλώσης καυσίμου αλλά απλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να επιβληθεί σε όλους παρά τη θέλησή του. Θα πρέπει η αγορά να το αποφασίσει. Αν θέλει ο κόσμος μετρητές, θα μπουν μετρητές και ενδεχομένως να έχει... Να θέλει ο κόσμος να πληρώσει και κάτι παραπάνω. Και πολύ φοβάμαι ότι η ομάδα μου είναι μετακίνητη στο θέμα αυτό. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να πείσουμε τις άλλες ομάδες, αλλά θα συνεχίσουμε να το πολεμάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάλτον. Σαφής η απόψη σας για αυτό το θέμα. Για την Άλντε, η κυρία Τσαράνσοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και αυτές τις προτάσεις. Δυστυχώς η ομάδα μου δεν μπορεί να τη στηρίξει όμως. Όπως ανέφερε και ο Ντάνιελ προηγουμένως, οι μετρητέ ε, κατανάλωση καυσίμων μπορεί να είναι χρήσιμοι μεν, αλλά το να είναι υποχρεωτικοί και να θεσπιστεί τέτοια υποχρέωση δημιουργεί πολύ σοβαρό άχθος. Το 6β εκτιμώντα ε, παραθέτει μια σειρά προβλημάτων. Έτοιμα μόνιμης ορατότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε εκ νέου ε, τους μετρητές που έχει καθένα στο αυτοκίνητό του για να φαίνεται και αυτή η μέτρηση. Το GPS πάντα θα πρέπει να δείχνει ε, αυτή τη μέτρηση ακόμα και όταν είναι απραργοποιημένο. Μετά, η προτινόμενη σύγκληση ό,τι αφορά την κατανάλωση που προβάλλεται και την πραγματική κατανάλωση. Δεν έχω καμία ιδέα πώς θα μπορούσε να οριστεί κάτι τέτοιο ή να διορθωθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα, ολο, ένα ολοκένουργιο ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο ε, για τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο θα ε, μετρούμε αυτά τα ποσά. Και τέλος, ο συμβιβασμός προσδιορίζει το FCM μόνο σε ό,τι αφορά το μετρικό σύστημα. Εγώ αφενός ε, πραγματικά θα ήθελα και το Ερμηνό Βασίλειο να υιοθετήσει το μετρικό σύστημα, όμως από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο οι ε, Βρετανοί θα τα κατανοήσουν όλα αυτά όταν βλέπουν χιλιόμετρα και όχι μίλια εν γέννη δεν με έχει πείσει επαρκώ η αξιολόγηση δικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη στηρίξω. Για την υπόλοιπη γνωμοδότηση, παραλαμβάνω την αντίρρησή μου σε ό,τι αφορά τη χρήση καταστάσεων πράξεων και να υπογραμμίσω ότι δεν θεωρώ ότι νέα πρότυπα εκπομπών θα πρέπει να τεθούν. Ευχαριστούμε. Πασκάλ Ντιουρόν, εξ ονόματος των Πρασίνων, θα μιλήσετε. Ακούστε, θα μιλήσω για τους πρασίνους πολύ σύντομα. Αρχικά βεβαίως ε, με μεγάλη χαρά ακούω την Ευελίνα όπως πάντα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα οικολογικά ζητήματα αποτέλεσε προτεραιότητα σε αυτό το εξαιρετικό κατά τα άλλα έργο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ. Προφανώς όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Συνεχώς ακούμε ότι προσπαθούμε να θέσουμε και να θεσπίσουμε κοινά πρότυπα για να μειωθεί η κατανάλωση και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του περιβάλλοντος, όμως ποτέ δεν, δεν ενσωματώνουμε όλο αυτό το ότι αν δεν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά και συνεχίσουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Συνεχώς λοιπόν αναφερόμαστε στο κόστος χωρίς να λάβουμε υπόψη τις προεκτάσεις μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό πλαίσιο. Πράγματι, τα οχήματα αυτά ε, ρηπαίνουν και πράγματι πρέπει να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό είναι υποχρέωση και για την δημόσια υγεία και για την οικονομία μα και την ευρωπαϊκή οικονομία εν γέννη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση να γίνει με μια ισορροπία μεταξύ κόστους και από τη μία πλευρά και από την άλλη όμως. Όχι μόνο να λέμε ότι πρέπει να γίνουν δαπάνες που θα προκύψουν από την ε, υποχρέωση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πράγματι υπάρχει κόστος εκεί για τα οχήματα και τους κινητήρες, αλλά στη Γαλλία βάση του ΠΟΗ, και δεν μιλώ για οικολογικό εδώ οργανισμό, αλλά για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ε, προκύπτουν λοιπόν 15.000 πρόοροι θάνατοι και πολλά προβλήματα υγείας εξαιτίας της ρήπανσης. Όλα αυτά εξαιτία των μικροσωματιδίων. Ήθελα λοιπόν να το επισημάνω αυτό ότι πρέπει να βρεθεί μια καλή ισορροπία. Αλλά όχι θα λύσουμε και αυτό το ζήτημα εδώ. Ευχαριστώ πολύ Βασκάλ. Επικαιροποιημένε μελέτε, οι έρευνε σίγουρα υπάρχουν για τι δαπάνε και για την ε, θέσπιση υποχρεωτικού συστήματο και για τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. σω κάποιο θα μπορούσε να τα αντισταθμίσει αυτά τα δύο. Ε, Νίκολα Ντάντι, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου, γιατί μια σειρά τροπολογιών που κατέθεσα εγώ για ε, την επισκευή έχουν ληφθεί υπόψη στην νομοδότηση. Για το μεθάνιο και άλλες ε, καλά και άλλα καύσιμα. Μειώνεται λοιπόν η κατανάλωση και η εκπομπή μάλλον μεθανίου... ό,τι φορά τη ρήπανση, όμως έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στη χώρα μου και αλλού για να καταφέρουμε να έχουμε ένα δίκτυο κατανομής του μεθανίου ως ε, τμήμα του συστήματος οχημάτων που είναι πολύ λιγότερο ρηπαίνων σε σχέση με ε, την τρέχουσα μορφή καυσίμων που αξιοποιείται. Και θα θέλαμε σε αυτή τη γνωμοδότηση να τονίσουμε την προετοιμασία μιας μέτρησης ε, του διοξιδίου του άνθρακα που μεταξύ μεθανίων και άλλων καυσίμων δεν μπορούσε να γίνει. Ξέρω ότι έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες που έχουν ληφθεί υπόψη και νομίζω ότι το μεθάνιο σίγουρα ρηπαίνει την ατμόσφαιρα όπως και άλλα καύσιμα, όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ του οχήματος που καταναλώνει καύσιμο και άλλου οχήματος που χρησιμοποιεί άλλο καύσιμο. Αυτό ισχύει σε πολλές χώρες και Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο κλίμα που να αλλάζει η ατμόσφαιρα με τη βροχή. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερως όταν έχουμε μακρόχρονες περιόδους ε, ξηρασίας και έτσι το μεθάνιο φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τα επίπεδα λοιπόν αυτά έχουν πέσει. Έχουμε μειώσει την χρήση μεθανίου και έχει δημιουργηθεί και ένα ε, δίκτυο κατανομής. έχει σταματήσει αυτή η προσπάθεια σύγκρισης μαθανίου με άλλα κάψιμα και αυτό είναι πολύ σωστό. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνεται και μια μέτρηση και τυποποίηση των μετρήσεων, όμως συνάδει και σύγκριση με άλλες μορφές καυσίμου. Ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό και να ληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στην Εβελίν. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, Πασκάλ δεν είναι μόνο οι πράσινοι αλλά και οι σοσιαλδημοκράτε αυτοί που θέλουν να έχουμε ένα υγιεινό περιβάλλον. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξή. Η ποιότητα τη ατμόσφαιρας και οι εκπομπέ. Ασφαλώ, συνδέονται και πάρα πολύ με την παραγωγή με την κατανάλωση ε, καυσίμων των αυτοκινήτων και διάφορες μελέτες καταδεικνύουν ότι αυτά που επισημαίνουν οι παραγωγή και αυτά που ισχύουν στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε ε, κοινέ μεθόδους καταμέτρησης για να υπάρχει συγκρισιμότητα. Για να μην ε, έχουμε αυταπάτες. Και κάτι άλλο το οποίο εμείς ως σοσιαλδημοκράτες ε, γενικά επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, όχι μόνο στον τομέα αυτό, όταν γίνονται μελετές τύπου. Να μην κοιτάμε μόνο τη μία πλευρά, αλλά να έχουμε μία συνολική προσέγγιση. Και εδώ θέλω να πω στον Πασκάλ το εξή, ότι φυσικά αν κάνουμε μελέτες αντικτύπου, το θέμα δεν είναι μόνο τι κοστίζει στις επιχειρήσεις, αλλά τι γίνεται στον τομέα της υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης, στην ε, επιδιόρθωση των περιβαλλοντικών καταστροφών, σε άλλους τομείς, ε, στο βιωτικό επίπεδο, στις καλύτερες συνθήκες ε, διαβίωσης του κόσμου. Όλα αυτά θα πρέπει να λεπτούν υπόψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαρκώς επαναλαμβάνουμε για τις μελέτες αντικτύπου. Δεν είναι δυνατόν να κοιτάμε μόνο μερός μόνο την οικονομική πτυχή. Θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά τι γίνεται. Και φυσικά πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για το φορολογούμενο, αλλά και να βελτιώσουμε τον τρόπο διαβίωσης τους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κύριε Γραπίνη έχει το λόγο. Ναι, θα είμαι σύντομη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς, ότι πάντα είναι πιο φθηνή και αποτελεσματική η πρόληψη από τη θεραπεία. Η πρόληψη λοιπόν, προστασία του περιβάλλοντος ως εκ τούτου, με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει χωρίς κόστος. Δεν κοστίζει τίποτα αν δεν εφαρμόσουμε αρκετά το σκέλος της πρόληψης, αυτό θα οδηγήσει σε ένα κόστος προκειμένου να αλλάξουν τα συστήματα, να αλλάξουν οι συνέπειες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τα θέματα της αποδοτικότητας, τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα τα οποία θα κληθούμε να αλλάξουμε, θα πρέπει να αλλάξουν τα συστήματά τους, η επένδυση λοιπόν για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτά Όλοι μαζί από κοινού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τη διάσταση αυτή. Από αριστερά, δεξιά, στο το κέντρο του πολιτικού φάσματος είναι καλύτερη η πρόληψη παρά η θεραπεία και όπως είπε και ο Πασκάλ, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές εδώ. Θα πρέπει πραγματικά να πετύχουμε ε, μια νέα ισορροπία. Δεν ξέρω ποιος έκανε την αξιολόγηση αυτή, αλλά όταν κάνει κανείς μία επένδυση, δεν κοιτάμε μόνο τα αριθμητικά στοιχεία, κοιτάμε τι θα γίνει και σε ένα βάθος χρόνου, σε 5, 10, 15 χρόνια, τι θα γίνει και πώς θα αποδώσει η επένδυση αυτή και κατά πόσον ε, μπορεί να έχει αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, Λίτρα. Θέλει κανείς άλλος να κάνει κάποια σχόλια. Εντάξει, θα έχουμε λοιπόν, ε, θα γίνει η ψηφοφορία για την ε, έκθεση αυτή στις 29 Ιουνίου για τις 15 Ιουλίου προβλέπεται ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, ΕΝΒΗ. Και μιας και δεν υπάρχουν ε, άλλα θέματα, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση κατά εξαίρεση πολύ πιο νωρίς. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι.